Dear colleagues. συνάδελφοι, σας χαιρετάω στο, στο σημερινό μας, σημερινή μας συνεδρίαση για να συζητήσουμε τις σχέσεις της, ε, της ε, Ευρωπαϊκής Ενώσεως και των Ηνωμένων Πολιτειών κατόπιν της ε, οικονομικής ε, και κοινωνικής κρίσεως και δεν ξέρω αν είναι το τέλος ε, ή είμαστε στη μέση και θα ήθελα να συζητήσουμε για τα θέματα που τίθενται και ποιες είναι οι προκλήσεις και έχουμε δύο ο επιφανείς ομιλητές που θα το συζητήσουν αυτό. Τι, αυτό, το δεύτερο, ε, τον ε, ε, πρόσωπο, τον κύριο Τζόζεφ Μέισον από τη Λουιζιάννα, Μπατόν ε, Ρούζ, ο επιφανής ε, καθηγητής στο Wharton School ε, Πανεπιστήμιο της Πενσιλβανίας και επίσης τον, τον κύριο Μπενουά Κερέ, ο οποίος είναι επιφανής προσωπικό οπότε ε, εφόσον έχουμε ήδη καθυστερήσει 10-15 ε, λεπτά πρέπει να ξεκινήσουμε αμέσως. Καταρχήν θα μιλήσει ο κύριος Μέισον και μετά ο Πίτερ Γιούγκερ, ο οποίος είναι πρόεδρος του Κέντρου Καπιταλισμού και Κοινωνίας στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια της Νέας Υόρκης. Ε, θα υπάρξει στην αρχή μία παρουσίαση και μετά, επειδή θα είναι δεκάλεπτη, εάν θεωρήσετε ότι χρειάζεται περισσότερο χρόνο, θα έχετε τη δυνατότητα να δευτερολογήσετε. Ο κύριος Μέισον, ευχαριστώ. Θα αναφερθώ και στους τέσσερις τομείς οι οποίοι αναφέρονται στην περίπτωση και θα ήθελα να αναφερθώ τώρα απαντώντας σε ερωτήσεις όταν θα μας επισκεφτείτε στη Washington. Καταρχήν δεν έχει τελειώσει η κρίση διότι υπάρχουν ακόμη πολλά δάνεια τα οποία δεν έχουν ρυθμιστεί στις Ηνωμένε Πολιτείες και υπάρχουν ε, ε, και ε, ορισμένα άλλα δάνεια τα οποία τώρα ναι μεν έχουν τύχει ένα διαπραγματεύσεως αλλά αυτά τα οποία έχουν υπομείνει της εποχής του 2006-2007 είναι τα ιδιαίτερως τοξικά και ε, θα μας απασχολήσουν για μία πενταετία και ε, υπόκεινται μεγάλες πιέσεις για να μπορέσουν να ρυθμιστούν. Έχουν γίνει προσπάθειες ε, για να καλυφθούν οι επενδυτές και οι ιδιοκτήτες ιδιοκτησιών αλλά δεν έχουμε μέχρι στιγμής επιτύχει και βλέπουμε ότι ε, υπάρχει μία αύξηση των CDS και ότι υπάρχει μεγαλύτερος κίνδυνος. Οπότε θα δείτε ε, ή στη διαφάνεια ότι ε, όλοι θέλουν να ισοσκελίσουν τον υπολογισμό τους χωρίς όμως οικονομίες και μια τέτοια δυνατότητα δεν είναι εφικτή στα πλαίσια του συστήματος. Αλλά ε, δημιουργείται όλο και μεγαλύτερη ασάφηση και μία λεπτομερής εξέταση του ΛΑΙΜΠΟΡ το 2007-2008 αποδεικνύουν ότι υπάρχει μειωμένη αποπληρωμή και ότι ουσιαστικά η κατάσταση έχει επιδεινωθεί. Γι' αυτό όπως γνωρίζετε ένα μεγάλο Μέρο μέρος οφείλεται εις ε, τα λάθη των Ηνωμένων Πολιτειών άρα μπορεί ε, οι λανθασμένες πολιτικές να δημιουργήσουν ένα κίνδυνο στο σύστημα. Τι είναι αυτό? Systemic risk. Ε, είχε εξεταστεί η κρίση κατόπιν της μεταδοτικής φύσεως της ασθενείας όπως εις το ανθρώπινο σώμα και μετέθεσε σε αυτή την παρομοίωση ή στο οικονομικό σύστημα ή στις διάφορες χώρες και ε, παρόλο που υπάρχουν πολλές σχέσεις ε, σε πολλαπλή, με πολλαπλές παθογένειες το θέμα εξαρτάται από τη συμπεριφορά του ανοσοποιητικού συστήματος οπότε ε, με την, με την ε, ε, με το θέμα αυτό πρέπει κανείς να συσχετίσει την ανεξαρτησία των εθνικών δημοσιονομικών συστημάτων. Οπότε πρέπει σαν λύση να μιλήσει κανείς ή για ακροτηριασμό ή για μεταμόσχευση και, ή για εμβολιασμό. Ε, ο ακροτηριασμός δεν είναι δυνατός. Ο ε, εμβολιασμός δεν είναι δυνατός διότι η κάθε κρίση έχει μοναδικά στοιχεία και άρα παραμένει το θέμα της μεταμόσχευσης. Πώς όμως μπορούμε ε, να μεταμοσχεύσουμε συστήματα τα οποία έχουν αποτύχει. Χρειάζεται πειθαρχία των αγορών Λοιπόν για να μπορέσουν να μειώσουν το βάρος το οποίο υφίστανται οι δημοσιονομικοί οργανισμοί για να μπορέσουν να ανεχθούν τα μοσχεύματα. Ε, γι' αυτό και θα πρέπει κανείς να αντιδράσει στην αγορά προτού φτάσει ο οργανισμός στην χρεοκοπία. Βεβαίως η έννοια αυτή ε, μας αποδεικνύει ότι δεν μιλάμε μόνο για ένα σύστημα ε, και θα πρέπει να έχουμε ήδη δράση προτού ο ένας ήδη ασθενής οργανισμός ε, μεταδώσει την ασθένεια και σε άλλους και ακόμη και σε δημοσιονομικές κρίσεις πρέπει να αντιληφθούμε ότι ε, ε, εάν πρόκειται για έναν μεγάλο οργανισμό θα μπορέσει ο οργανισμός αυτός να διαιωνιστεί επαόριστον χωρίς, ε, θέτοντας σε κίνδυνο τις επόμενες μονάδες για την επόμενη κρίση και υπάρχει όντως ένα πρόβλημα και πρέπει να να μειώσουμε τον ε, συστηματικό κίνδυνο ε, διότι ε, ε, πρέπει ε, κανείς ε, να εξετάσει την ασφάλεια από τους οργανισμούς οι οποίοι εποφελούνται της στηρίξεως της κυβερνήσεως διότι θα πρέπει να υπάρξει πειθαρχία στην αγορά για να αποφευθεί η στήριξη από το κυβερνητικό σύστημα. Πρέπει να δούμε εάν η βοήθεια ε, πρέπει ε, να ληφθεί εντός του συστήματος ή εκτός του συστήματος. Δηλαδή, ε, εάν ε, περιμένει κανείς ε, να φτάσει στη χρεοκοπία ε, μία, ένας οργανισμός οι επενδυτές θα δυσπιστήσουν προς ολόκληρο το σύστημα. Άρα ο νομοθέτης θα πρέπει να έχει λύσει το πρόβλημα προτού το αυτό επιδεινωθεί και δεν πρέπει να νομοθετούν μόνο αλλά θα πρέπει να παρακολουθούν και τις αγορές οι οποίες ακόμη είναι και εκτός του νομοθετικού πλαισίου ώστε ε, να αξιολογούν τον κίνδυνο ο οποίος ε, φτάνει στο μετέχμιο διότι διαφορετικά θα έχουμε ένα δημοσιονομικό πρόβλημα το οποίο θα είναι συστηματικό ενώ με τον περιορισμό αυτό αυτό μπορεί να υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα αλλά δεν θα επηρεάσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών. Τι πρέπει λοιπόν να γίνει. Καταρχήν πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι το διεθνές σύστημα είναι ευάλωτο από οικονομικά σοκ και το βασικό είναι ε, να εξετάσει κανείς τις γωνίες προς δεξιά και αριστερά διότι η στα αριστερά υπήρχε μία, ένας μικρός κίνδυνος ενώ δεξιά μετά από το, την μεγάλη κρίση υπάρχει μεγάλος κίνδυνος άρα έχουμε ακόμη πολύ δρόμο μπροστά μας και ε, παρόλο που ε, ε, ε, λαμβάνονται μέτρα ορισμένες χώρες αντιμετωπίζουν δημοσιονομικά οικονομικά προβλήματα και φορολογικά προβλήματα και βλέπουμε ότι ε, τελικά ο προπολογισμός των Ηνωμένων Πολιτειών είναι ο τέταρτος χειρότερος ε, μετά την ε, Ισπανία, την Ταϊλάνδη και κάποιες άλλες χώρες και χειρότερος από της Ελλάδος και άλλων χωρών. Βλέπουμε λοιπόν ότι όλα αυτά τα θέματα έχουν δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα μπορούμε να δημιουργήσουμε μία περαιτέρω φούσκα αλλά αυτό δεν θα μας λύσει το πρόβλημά μας και ε, χρειάζεται μία οργάνωση η οποία θα δημιουργήσει οικονομική αξία και ανάπτυξη αλλά τα χρήματα απλώς δεν μπορούν να επανακτήσουν την εμπιστοσύνη των επενδυτών ούτε να δημιουργήσουν ανάπτυξη. Πρέπει να υποκινήσουμε την ε, ανάπτυξη ή να περιμένουμε να υποχρεωθούμε όπως έγινε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Τέλος, καταλήγοντας θα ήθελα να πω ότι κανένα από τα θέματα δεν είναι νέο διότι ε, τα προβλήματα αυτά διαιωνίζονται εδώ και 40 χρόνια περίπου. Χρειάζεται ένα μόνιμο πλαίσιο στο οποίο να ενταχθούν οι ε, μεταρρυθμίσεις. Δεν χρειαζόμαστε έναν ειδικευμένο οργανισμό αλλά θα πρέπει να προσπαθήσουμε ε, να προχωρήσουμε σταθερά και αργά ε, προς ε, την θεσμική διαιτησία και ελπίζουμε ότι κατά αυτόν τον τρόπο θα προλάβουμε την επόμενη κρίση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα θα προχωρήσουμε στον επόμενο ομιλητή και μετά θα ξεκινήσει η περίοδος των ερωταπαντήσεων. Άρα δίνω το λόγο στον επόμενο ομιλητή. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Στην Ευρώπη υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που πιστεύουν ότι αν δεν είχαμε την κρίση και την κατάρρευση της ε, Λίμαν, δεν θα είχαμε αυτή την κρίση. Αυτό είναι λάθος. Και θεωρούν ότι το λάθος της ε, Αμερικανικής κυβέρνησης είναι ότι διέσωσε την ε, Λίμαν, αλλά το έκανε πολύ καθυστερημένα. Αν είχε, δεν είχε περιμένει τόσο πολύ, η κρίση θα ήταν λιγότερο σοβαρή. Ε, τα τελευταία χρόνια είχαμε μια τεράστια ανάπτυξη από 23 ε, τρισεκατομμύρια δολάρια σε 58 τρισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίω. Ποτέ δεν είχαμε τέτοια ανάπτυξη. Ε, στο παρελθόν είχαμε και άλλες κρίσεις. Ο καπιταλισμός διέπεται από κρίσεις. Αλλά το θέμα είναι πόσο αποτελεσματικό είναι, πόσε γνώσει γνώσεις εμπεριέχει, πόσο δυναμική είναι η οικονομία, ε, ούτως ή άλλως ε, υπάρχουν, ε, υπάρχουν κρίσεις. Η, πρώτη τελευταία ήταν του 29. Χωρίς την κρίση η φούσκα και ειδικά η φούσκα των ακινήτων θα ήταν πολύ μεγαλύτερη και θα ήταν πολύ πιο δύσκολο να την περιορίσουμε και να τη διορθώσουμε. Η Ούτως ή άλλως θα είχαμε αυτές τις διαταραχές ε, ε, και παγκόσμια και στην Ευρώπη και παρότι έχουμε και τώρα δυσκολίες θα ήταν πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα αν δεν υπήρχε αυτή η φούσκα. Ε, αν πιστεύουμε τώρα ότι είναι δύσκολο να επιλύσουμε το πρόβλημα, φανταστείτε τι θα γινόταν αν οι φούσκες μεγάλωναν ακόμα περισσότερο, το πρόβλημα θα διωγγωνόταν και το τέρας θα μεγάλωνε ακόμα περισσότερο και θα μπορούσαμε να το αντιμετωπίσουμε. Οι παγκόσμιες αυτές ανισορροπίες ε, αύξηση του όγκου του χρήματος, ε, το παγκόσμιο χρέος, ε, οι στεγαστικές πολιτικές στις Ηνωμένε Πολιτείε όντως ήταν απαράδεκτες. Παραδείγματος χάρη κάποιος παίρνει υπόθεκο δάνειο 700.000 δολαρίων ενώ δεν έχει εισόδημα, ενώ δεν έχει ένα χαρτοφυλάκιο αξιογράφων. Πώς θα μπορέσει να αποπληρώσει αυτό το χρέο. Επομένω, δεν λειτουργήσε το σύστημα, δεν λειτουργήσαν οι ρυθμίσει για τι ε, για τράπεζες. Ορισμένοι λένε θέλουμε περισσότερες ρυθμίσεις ή καλύτερε ρυθμίσει. Για... Το θέμα είναι, πριν βγούμε από αυτή την κρίση, το θέμα είναι να καταλάβουμε πώς μπήκαμε σε αυτή την κρίση. Ε, στην Ευρώπη μιλάμε πάρα πολύ για τις ρυθμίσεις εμείς στι ΗΠΑ μιλάμε περισσότερο για τη δομή. Για δομικά θέματα. Παραδείγματο χάρη, δύο μέρε πριν ανακοινώσει ο πρόεδρο Ομπάμα τον κανόνα, ε, το μέτρο Βόλκερ, και ένα δεν ήξερε τίποτα. Ορισμένοι λένε ότι θέλουν να περάσει στην ιστορία τουλάχιστον με ένα τέτοιο σχέδιο για τον πρόεδρο Ομπάμα. Ε, έχουμε ρυθμίσει με λάθος τρόπο τα λάθος πράγματα και τώρα εστιάζουμε πάλι λάθος, σε λάθος πράγματα ε, στις εμπορικές τράπεζες. Σε εμπορικές τράπεζες που ε, το παίζουν επενδυτικές τράπεζες, ενώ δεν είναι επενδυτικές τράπεζες. Ε, δεν είδαμε όμως το πρόβλημα με τα hedge funds και με τα private equities η μέση μόχλευση στην τράπεζα ήταν 30-40 στις ΗΠΑ, ενώ ε, στην Ευρώπη ήταν 40 με 50. Ενώ στα, η μέση μόχλευση ε, στα hedge funds ήταν 3 με 4. 1 προς 10 δηλαδή. Έχουμε επίσης πολλές ανισορροπίες, πολλές ανισόρροπες δραστηριότητες. Παραδείγματος χάρη, το, το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, αυτό προσπαθεί να ρυθμίσει τις ανισορροπίες. αλλά δεν ούτε στο χρέος καμίας κυβέρνηση, ούτε στο χρέος Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, στην πραγματικότητα είναι 7 φορές το, ο προπολογισμό Ευρωπαϊκής Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένω, ε, οδηγούμε την Ευρωπαϊκή Ένωση σε αφαιρεγγιότητα. Δημιουργούμε όλες τις προϋποθέσεις για ανισορροπίες. Οι εταιρείε βαθμονόμησης της πιστοληπτικής ικανότητας έδωσαν 3α σε 66.000 προϊόντα. Οι εταιρείε αυτές έχουν, λειτουργούν με πολύ λαθασμένο τρόπο. Θα μπορούσαμε να τις καταργήσουμε. Ούτως ή δεν έχουν κανόνες, δεν είναι αποτελεσματικές, μας παραπλανούν και στην πραγματικότητα τους πληρώνουν οι επενδυτές, αλλά οι εκδότες ούτως ή άλλως. Παραδείγματο χάρη. Ε, εσείς ας πούμε, αν εγώ θέλω να πουλήσω ένα σπίτι και εσείς θέλετε να το αγοράσετε ας πούμε ε, και επιβάλλω μία τιμή με βάση μόνο τα δικά μου ε, στοιχεία, αυτό είναι τελείως λάθος. Οποτεδήποτε ανεβα... ανεβάζει τη βαθμολογία η εταιρεία, συνήθω είναι... έχει λάθο. Επίσης, η βασιλεία είναι λαθασμένη έννοια. Υπάρχει λιγότερη μόχλευση αν θες να επενδύσεις σε ένα υπόθηκο δάνειο. Και αν επενδύσει σε CDO, υπάρχει μια προϋπόθεση για equity. Αν διαβάσατε το βιβλίο του Μάικ Λούις, θέτει το ερώτημα ποιος θα αγοράσει, θα αγοράσει τα CDOs. Στην Ευρώπη Είχαμε αυτή την κρίση επίσης στην επενδυτική κρίση οι Ευρωπαίοι επενδύουν περισσότερο από τους Αμερικανούς. Ο Λουίς ε, θέτει το ερώτημα ποιος αγοράζει όλα αυτά τα πράγματα και κάποιος ψιθυρίζει τον Ντίσεντολφ, οι ανόητοι Γερμανοί. Ε, το Ντίσεντολφ είναι η IKB. Στη μόνη χώρα όπου η, η κυβέρνηση δεν μπορούσε να γλιτώσει τις ε, προβληματικές τράπεζες ήταν η Γερμανία, γιατί ούτως ή άλλως ήταν ιδιοκτήτης των τραπεζών αυτών. Η Ευρώπη λοιπόν ε, θα δυσκολευτεί πάρα πολύ να αντιμετωπίσει το πρόβλημά της. πρόκειται όταν δυσκολευόμαστε να βγούμε από την κρίση, ε, λέμε ότι το πρόβλημα είναι πολιτικό και οικονομικό. Αυτό είναι σαν Το πρόβλημα είναι χρηματοπιστωτικό. Η παγκόσμια οικονομία κάθε χρόνο δημιουργούσε 42 εκατομμύρια θέσεις εργασίας. Κάθε χρόνο. και χάσαμε πολύ λιγότερα από αυτά που δημιουργήθηκαν. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να πληρώσουμε το τίμημα. Οι Ευρωπαίοι αντιμετωπίζουν ε, με πολύ διαφορετικό τρόπο την κρίση. Η ΕΚΤ αγοράζει τώρα ομόλογα. Όχι από τις ε, κυβερνήσεις απευθείας, αλλά από τις τράπεζες. Στην πραγματικότητα όλο αυτό το πρόγραμμα είχε σαν σκοπό να διασωθούν οι τράπεζες. Ε, μπορείτε να δείτε τον κατάλογο των ελληνικών ομολόγων, ε, ποιος τα έχει αυτά τα ελληνικά ομόλογα. Στην πραγματικότητα αγοράζουν ελληνικά ομόλογα. Γιατί τα αγοράζουν. Αυτά τα ομόλογα αξίζουν 20, 25 δισεκατομμύρια συγγνώμη, ευρώ από τα 700 τόσα. Οι κυβερνήσει λένε ότι πρέπει να κάνουμε τα πάντα για να υπερασπιστούμε το ευρώ. Στρατηγικέ εξόδου, αλλαγέ αλλαγές στην Ελλάδα. Η Ελλάδα δεν θα μπορέσει ποτέ να πληρώσει αυτά τα λεφτά. Ε, όποιος σας λέει το αντίθετο ψεύδεται. ούτως ή άλλως ε, ο λόγος χρέους προς ΑΕΠ θα πάει στο 150% όσον ούπο. Και οι υπόλοιπε χώρες αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα. Για πρώτη φορά είδαμε ότι το CDS για τις 15 παλιές χώρες είναι μεγαλύτερο από τις μεγάλες ευρωπαϊκές εταιρείες. Επομένως, οι αγορέ ε, εκτιμούν ότι υπάρχει μεγάλη περίπτωση χρεοκοπίας μίας από τις 15 παλιέ ευρωπαϊκές χώρες. Για να κλείσω με, αυτό το, με τα σχόλια περί τραπεζών, αυτό που χρειαζόμαστε είναι μια πλήρη συζήτηση για το, τη διάρθρωση του τραπεζικού τομέα. Αναθεώρηση των ρυθμιστικών κανόνων. Μέχρι στιγμή στην Ευρώπη δεν υπήρχε τίποτα και μεταρρύθμιση των ε, rating agencies, ε, μεταρρύθμιση της Βασιλείας. Πολλές ε, δημόσιες τράπεζες κάναν λάθη, λάθη που δεν έκαναν όλες οι ιδιωτικές τράπεζες. Η απαγόρευση του short selling είναι σαχλαμάρες. Το, αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι είναι το πολύ πολύ ουδέτερο το short selling. Ε, κοιτάξτε το κείμενο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, σελίδες 49 με 53, ε, που λένε μην το αγγίξετε το short selling, θα καταστρέψει αγορές αν το αγγίξετε. Θα κάνουμε τη συζήτηση για τις δομές, για την αρχιτεκτονική. Ούτως ή άλλω ε, θα συζητηθεί και το σχέδιο Βόλκερ, όχι, και ούτως ή άλλω δεν θα πρόκειται να εφαρμοστεί με τον απλό και καθαρό τρόπο που θα ήθελε ο ίδιος. Λίγες παρατηρήσεις τώρα για το πώς μπορούμε να ξεπεράσουμε το πρόβλημα και μέσω ποιου πράγματος, ε, μέσω της ενίσχυσης της απασχόλησης και της τόνωσης της πραγματικής οικονομίας. Ε, η τόνωση δεν είναι ο τρόπος για να ξεφύγουμε. Δεν θεωρώ ότι είναι λάθος η ερώτηση, αλλά η τόνωση δεν λύνει το πρόβλημα. Ε, αναστήσαμε το Mark τον Keynes για 18 μήνες και τώρα ξαναπέθανε πάλι. Το αναστήσαμε αλλά πρέπει να πεθάνει, γιατί αποδείχθηκε ότι πηγαίνει προς τη λάθος κατεύθυνση. Δεν μπορούμε ούτως ή άλλως να συνεχίσουμε με, τα, με την αύξηση των δημοσίων δαπανών. Ούτως ή άλλως θα πρέπει να, να τα πληρώσουμε αυτά. Δαπανούμε και μετά πληρώνουμε. Η Ευρώπη θα πρέπει να ξεφύγουν από τις πολιτικές τους. Ε, θεωρείτε ότι η κυβέρνηση είναι φίλη σας μόνο αν πληρεί δύο προϋποθέσεις. Αν είναι μεγάλη και αν είναι αναποτελεσματική. Και ούτω ή άλλω και εσεί, αν είσαστε μεγάλο και αναποτελεσματικό, σα προστατεύει. Αν είσαστε μικρό και αποτελεσματικό, σα παρατάει. Ο μόνο τρόπο είναι μέσω τη καινοτομία. Μέσω τη επιχειρηματικότητα, μέσω τη δημιουργία δυναμισμού, μέσω νέων προϊόντων, νέων υπηρεσιών και νέων θέσεων απασχόληση για ανθρώπου που μέχρι στιγμή δεν είχαν απασχόληση. Δεν αντιλαμβανόμαστε σωστά ε, την ε, καινοτομία στην Ευρώπη. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τι είναι ε, εφεύρεση και τι είναι κοινοτομία. Ε, στην ε, εφεύρεση τα χρήματα γίνονται γνώση. Το αντίθετο είναι κοινοτομία. Τα λεφτά να τα κάνουμε γνώση, το κάνουμε καλά στην Ευρώπη. Αλλά τη γνώση να την κάνουμε λεφτά στην Ευρώπη, δεν ξέρουμε να το κάνουμε και εκεί θα πρέπει να βελτιωθούμε. Ο μόνος τρόπος για να ξεφύγουμε λοιπόν είναι αυτός, όχι μόνο. Το καλό είναι ότι η παγκόσμια οικονομία είναι πολύ καλύτερη, τα πάει πολύ καλύτερα από την ευρωπαϊκή οικονομία. Οι αναδυόμενες αγορές για πρώτη φορά ε, αποτελούν το 50% του παγκόσμιου ΑΕΠ. Τα τελευταία δέκα χρόνια η αύξηση του ΑΕΠ ε, προήλθε κυρίως από τις ε, αναδυόμενες οικονομίες και κυρίως από τις BRICS. Οι αναδυόμενες αγορές αποσυνδέονται από τα προβλήματά μας και εμείς πρέπει να συνδεθούμε με το τι συμβαίνει σε αυτές τις χώρες. Κοιτάξτε την Κίνα. Πριν από 10 χρόνια η συνεισφορά της Κίνας ε, στο παγκόσμιο ΑΕΠ ήταν το 17%. Τώρα, ε, την επόμενη χρονιά θα φτάσει ενδεχομένως στο 30%. Αυτό θα είναι θετικό και για την Ευρώπη και για κάποιες από τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν πολλά προβλήματα. Για το ευρώ να πω δύο λόγια. Δεν πρέπει να ντρεπόμαστε που το ευρώ είναι 1,22. 1,22, 1,23, αλλάζει, ούτως ή άλλως παίζει. 7 χρόνια υπάρχει, 8 χρόνια. Τα περισσότερα ήταν πάνω από 1,25. Η Goldman Sachs έκανε ένα υπολογισμό της προάλλης και το δημοσίευσε. Και είπε ότι η πραγματική τιμή είναι μάλλον γύρω στο 1,22. Δεν είναι άσχημα. Τώρα εστιάζουμε το πρόβλημά μας στον Ευρωπαίο καταναλωτή. Ε, βλέπετε τα διάφορα προβλήματα που έχει η ευρωπαϊκή οικονομία χάλιβα, ε, το βάρος που έχει ο Ευρωπαίος καταναλωτής λόγω των τιμών της ενέργειας και του πετρελαίου. Ούτως ή άλλως η ευρωπαϊκή ε, βιομηχανία χάλιβα είναι πάνω από το 30% τώρα. η δυνατότητα ε, πλεονάσματος της ε, βιομηχανίας χάλιβας στην Κίνα είναι ακόμα μεγαλύτερη. Η παραγωγή, η κινέζικη παραγωγή ε, χάλιβα είναι πολύ μεγαλύτερη από τη συνολική ευρωπαϊκή παραγωγή. Ούτως ή άλλως δεν παράγουμε στο 100%, 100 του δυναμικού μας. Εμείς δημιουργούμε τις ανισορροπίες. Πολύ περισσότερο από το κάνουμε στο παρελθόν. Το 60% του κινέζικου χάλιβα εξάγεται στην Ευρώπη και στην Αμερική, σε ευρωπαϊκές και αμερικανικές εταιρείες. Εμείς δημιουργούμε τα πλεονάσματα των Κινέζων, τα έλλειμματα δικά μας. Πάντω σήμερα η παγκόσμια οικονομία είναι σε καλύτερη κατάσταση από ό,τι ήταν μετά την κρίση στη δεκαετία του 30. Γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι ζουν σε καπιταλιστικέ ε, οικονομίε, σε οικονομίε τη αγορά. Και υπάρχει φοβερό δυναμικό μείωση τη φτώχεια σε φτωχέ χώρε, ε, Ινδία, Κίνα, ακόμα και στην Αφρική. Και αυτό θα μα βοηθήσει για να ξεφύγουμε από την κρίση. Την εποχή που έγινε η κρίση ε, στη δεκαετία του 30, ο καπιταλισμό και η οικονομία τη αγορά ήταν πολύ μικρή. Ο περισσότερος πληθυσμός ζούσε σε άλλου τύπου συστήματα. Για να τελειώσω αισιόδοξα. Το πρόβλημα δεν είναι ότι εμείς συνεισφέρουμε, δηλαδή οι Ευρωπαίοι συνεισφέρουν για να ξεφύγουμε από την κρίση. Ούτως ή άλλως θα μας βοηθήσουν οι ανδιόμενες αγορές, αν δεν κάνουμε πολλά λάθη. Ευχαριστώ. Σε ευχαριστούμε πολύ. Περνάμε τώρα στις που Προτείνω στον πρώτο γύρο να ακολουθήσουμε τι πολιτικές ομάδε. Ποιο θα ήθελε να θέσει μια ερώτηση για του συντηρητικού παρακαλώ. Εσείς. Πολύ καλά. Εσείς. σα ευχαριστώ πολύ για τις δύο αυτές εισηγήσει σας. Είναι πολύ ενδιαφέρουσες ήταν. Μία ερώτηση θα ήθελα να διατυπώσω. Ίσως και στους δυο σα. Α ξεκινήσω όμω με τον κύριο Γιούγκεν. Να προσπαθήσω να το επικεντρώσω με οξυμένο τρόπο. Είπατε ότι η διέξοδος είναι η καινοτομία, ο δυναμισμό, νέε θέσει απασχόληση. Εξαιρετικό ακούγεται αυτό. Ω πολιτικό άνδρας επαναλαμβάνω αυτού του όρου αυτέ τι λέξει και είμαι σίγουρο και οι συνάδελφοί μου το κάνουν. Το πρόβλημα είναι ότι κανένα δεν φαίνεται να κατανοεί ακριβώ πώ αυτοί οι όροι, αυτέ οι λέξει θα αποκτήσουν ισχύ και αποτέλεσμα. Δεν φαίνεται από πλευρά των πολιτικών κάποιο να ήταν αντίθετο. Και είμαι βέβαιο ότι όλοι θα συμφωνούσαν ολόθερμα. Το ερώτημα όμω είναι ποια πολιτική απόφαση και ποιες πολιτικές αποφάσεις πρέπει να ληφθούν από την Ευρώπη που θα καταστήσουν εφικτή αυτή την εξέλιξη. Και η ερώτηση σε εσά θα ήταν πώς βλέπετε εσείς, δηλαδή τι πρέπει να γίνει από πλευράς πολιτικής χάραξης και νομοθετικής πρωτοβουλίας για να μπορέσουμε να, διέ, να διέλθουμε, να εξέλθουμε από αυτή την κρίση. Και σε σχέση με τις αντιδράσεις είναι όμω ε, γενικά αυτά και θα ήθελα να ακούσω την άποψή σα Ποια θα ήταν η δική σα συνταγή για τη διέξοδο από την κρίση. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ. Χαίρομαι πολύ που θέσατε αυτήν την ερώτηση, διότι φυσικά δεν μπορούσα να επισέθω σε λεπτομέρειε και πιο πριν. Α ξεκινήσω, αν επιτρέπετε, με το τι χρειάζεται η Ευρώπη. Η Ευρώπη χρειάζεται πιθανότατα πρόσθετα 6 εκατομμύρια επιχειρηματίε επιπλέον. Το πρώτο ερώτημα είναι πώ θα το καταφέρουμε να, έχουμε, να πείσουμε 6 εκατομμύρια παραπάνω πολίτε να ξεκινήσουν μια επιχείρηση και να γίνουν επιχειρηματίε. Πρέπει να του πείσουμε πρώτον ότι δεν θεωρούμε ότι είναι οι εχθροί μα. Δεν του θεωρούμε εχθρού. Δεν θεωρούμε ότι αυτοί είναι εκμεταλλευτέ που εκμεταλλεύονται άλλου ανθρώπου μέσω των δικών του πρωτοβουλειών. Πρέπει να το κάνουμε αυτό κατανοητό, να το κατανοήσουν οι πολίτε αν θέλουμε να κινηθούν προ αυτή την κατεύθυνση. Ότι δηλαδή πιθανότατα ως, ε, αν δεν το καταφέρουμε αυτό θα υπάρξει αποτυχία τρει, τέσσερι, πέντε σε σχέση με τα πρώτα πέντε χρόνια. Όχι μόνο χρειαζόμαστε ένα πολιτισμικό πλαίσιο εκείνων που κερδίζουν όπως και στην, στον αθλητισμό, αλλά και τι θα κάνουμε με εκείνου που αποτυγχάνουν. Χρειαζόμαστε ένα πολιτικό, πολιτισμικό περίγυρο για να ε, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε και τις αποτυχίες. Πρέπει να ενθαρρύνουμε λοιπόν τους πολίτες μας να ξεκινήσουν τέτοιες πρωτοβουλίες. Πρέπει να δημιουργήσουμε τη δημόσια εικόνα και οι πολιτικοί στην Ευρώπη έχουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο να διαδραματίσουν. Πρέπει να πούμε ότι ένας επιχειρηματίας είναι κοινωνικός ήρωας. Γιατί? Διότι υπομίζεται προσωπικά και οικονομικά και κοινωνικά κινδύνους για όσους απασχολεί. Τουλάχιστον λοιπόν μπορούμε να πούμε για όσους ε, απασχολούνται από αυτόν σε ένα χρονικό διάστημα. Πρέπει λοιπόν να έχουμε την ιδέα του ήρωα, όχι μόνο και της επιτυχίας στον αθλητισμό ή σε άλλα πλαίσια, αλλά πρέπει αυτό να υπάρχει και στο επιχειρήν, στους επιχειρηματίες. Δεν, είμαστε, δεν είμαι υπέρ τεράστιων αμοιβών για τους επιχειρηματίες. Είναι όμως μια λάθος συζήτηση σε μια χώρα, ας το πούμε στη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης, που θεωρούν οι πολίτες ότι είναι πραγματικά εξοργιστικό ο διευθύνων σύμβουλος ε, μιας τράπεζας να, ε, να παίρνει 11 εκατομμύρια ευρώ ετήσια. Ένας από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές της Bayern München παίρνει και αυτός 11 εκατομμύρια ευρώ. Όλοι όμως συμφωνούν με αυτό το μισθό. Γιατί συμφωνούν με αυτό οι πολίτες ενώ διαφωνούν για τον ε, εκτελεστικό μιας τράπεζας προφόρων 11 εκατομμύρια. Ενώ για τον αθλητή, τον αυτόν τον ποδοσφαιριστή είναι 11 εκατομμύρια μετά από την αγγλιστή ε, ε, παρακράση των φόρων. Η δεύτερη παρατήρηση που θα ήθελα να κάνω είναι ότι όχι μόνο δεν έχουμε αρκετούς ιδρυτές ε, επιχειρήσεων, έχουμε και έλλειψη αγγέλων επιχειρηματιών. Έχουμε έλλειψη πολιτισμικού περίγυρου εκείνων που θα υποστηρίζουν και θα τονώνουν την, το επιχειρήν και τους επιχειρηματίες και την τεχνογνωσία για την ίδρυση μιας νέας επιχείρησης η δυνατότητα αυτή δεν είναι παρά η μετάδοση, η μεταλαμπάδευση της τεχνογνωσίας και της ικανότητας από μια γενεά προς την άλλη. Αυτό χρειαζόμαστε. Έχουμε μια μη λειτουργούσα, θα έλεγα, μορφή του καπιταλισμού κινδύνου. Χρειάζεται το επιχειρήν με την έννοια του επιχειρηματικού κινδύνου δεν θα πρέπει εδώ να βασιζόμαστε σε πιστώσεις αλλά στο πού θα επικεντρώνονται οι ε, επενδύσεις. Εδώ υπάρχει ένα έλλειμμα το οποίο πρέπει να καλύψουμε και με αποτελεσματικό τρόπο. Τέταρτον, έχουμε έλλειψη κεφαλαίου κινδύνου. Το χρειαζόμαστε για τις επενδύσεις ε, σε ε, ταχεία, πω δόμηση, διάρθρωση νέων επιχειρήσεων. Κάποιοι πολιτικοί θεωρούν ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις πρέπει να μείνουν μικρών διαστάσεων για να μπορούν ε, να τις ε, υποστηρίζουν και να τις ε, τονώνουν οι πολιτικοί. Όμως πρέπει να καταστεί δυνατόν να ξεκινήσουν επιχειρήσεις και όχι μόνο να μείνουν μικρές αλλά να ταχύτατα να μεγεθυνθούν. Αυτό είναι σημαντικό. Και πέμπτον, σε στις έχουμε 3,6% ετήσια, δηλαδή 6 εκατομμύρια που ξεκινούν ετήσια σε σχέση με το ΑΕΠΑ έχουμε μικρό ποσοστό στην Ευρώπη. 75% όλου του κεφαλαίου κινδύνου είναι τον ΙΠΑ παγκόσμια. 18 δις ε, ε, ε, δολάρια πέρσι, συν επιπλέον 17 35. Αν τα προσθέσετε αυτά και δείτε τι γίνεται στην Ευρώπη, το πολύ πολύ 3,5 είναι η επίδοση της Ευρώπης. Στην Silicon Valley έχουμε 2,5 φορές σε σχέση με τις επενδύσεις στο ανθρώπινο δυναμικό ετήσια οι επενδύσεις στο ανθρώπινο δυναμικό 100% είναι. η επικεφαλής είναι το Ισραήλ με 250 με 10 ε, δολάρια ανακεφαλήν είναι, έχουμε την επίδοση των ΗΠΑ, 5 είναι η επίδοση της Ευρώπης ε, ανακεφαλήν, 5 δολάρια. Πρέπει εξειδικευμένα μέτρα να λαμβάνονται και ρυθμιστικά αλλά και στο φορολογικό σύστημα. Αν, μια τελευταία λέξη, αν έχετε φορολογία όπως στην γερμανική οικονομία, εκείνος που θα ξεκινάει μια επιχείρηση, startup, που είναι η μεγαλύτερη ε, επένδυση κινδύνου, φορολογικά θα ήταν το ίδιο σαν αγόραζε κανείς ε, ομόλογα της γερμανικής κυβέρνησης. Ε, λοιπόν, δώστε μας μια ευκαιρία να μπορέσουμε να το περάσουμε αυτό γιατί και να μην μείνουμε σε ένα παράλογο πλαίσιο σε σχέση με το κεφάλαιο κινδύνου για την ε, ε, τόνωση νέων επιχειρήσεων. Χάνουν τις, τα κεφάλαια αυτά μετά στη συνέχεια πλήρως. Υπάρχουν πολλά που μπορεί να κάνει κανείς ως πολιτικός λοιπόν βλέπετε. Ευχαριστώ. Πολύ σύντομα για κάποιες ε, για δύο πτυχές. Πρώτα απ' όλα συμφωνώ με τον κύριο Γιούγκεν για τον πολιτισμό των ε, νικητών, ε, εκείνων που κερδίζουν το παιχνίδι. Είναι πολύ σημαντικό για την δυναμική του συστήματός μας. Πρέπει να ενστερνιστούμε αυτό. Έχουν, τους αποκαλούμε πολλές φορές εκείνους που δεν πάνε καλά ως χαμένους ή εκείνους που χρεώνονται την αποτυχία, αποτυχημένους. Όμως πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Έχουμε αγώνα στη ΣΥΠΑ σε σχέση με την μεταρρύθμιση του πακέτου, νομοθετικού πακέτου για την ε, ανακούφιση των ε, ε, μέτρων που στις επενδυτικές πολιτικές δημιούργησαν δυσκολίες. Πρέπει να δούμε το πώς μπορεί να αντληθεί πρόσθετη αξία σε σχέση με αυτές τις επιχειρήσεις. Είναι ένα δύσκολο εγχείρημα σε σχέση με την μεταβατική περίοδο για το τις συμβάσεις ε, και το δυναμικό που αναπτύσσει ένας ε, ε, μικρομεσαίος επιχειρηματίας και να δούμε εδώ πώς είναι δυνατόν να μην παρεκκλίνει περισσότερο από τις πρακτικές μέσα στο, στον κύκλο εργασιών του. Πρέπει να αναγνωρίσουμε λοιπόν σε σχέση με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και την προοπτική για αυτές και ο κύριος Ιούγεν το επιβεβαίωσε αυτό για μένα πιο πριν η αποτυχία δεν είναι αποτυχία είναι κάτι το οποίο μας βοηθά να μάθουμε μάθουμε καλύτερα κάτι άλλο και να είμαστε καλύτεροι την επόμενη φορά που το αποτολμούμε και ξεκινάμε κάτι άλλο. Πρέπει με αυτόν τον τρόπο να δράσουμε και στο πολιτισμικό επίπεδο να υπάρξει η ιδέα ότι ο πολιτισμός του επιχειρήν είναι σημαντική υπόθεση. Να ξεκινήσει μια πολιτισμική, ας το πω έτσι, τόνωση για να υπάρξει ε, επενδυτική προσπάθεια και μπορεί κανείς σε σχέση με πολύ μικρότερο, μικρότερες ανεπτυγμένες χώρες να δει ότι υπάρχει ανθούσα ε, κοινωνική προσπάθεια όσον αφορά τις ε, πρωτοβουλίες στο επίπεδο των ε, επιχειρηματιών. Ακόμα και σε θα έλεγα ρηπαρές εργασίες που άλλοι θα τις απέφευγαν. Και έτσι υπό την προοπτική που εξετάζει κανείς αυτό και πολιτικά θέτεται το ερώτημα που διατυπώνουν πολλές ε, ε, αναπτυσσόμενες χώρες. Πού βρίσκονται οι ευκαιρίες για μας ε, ως χώρα τι είναι εκείνο το οποίο σε σχέση με το σύστημα παιδείας και εκπαίδευσης μπορεί να γίνει για να υποστηρίξει την ανάπτυξη σε διάφορες βιομηχανίες και βιομηχανικούς κύκλους ε, και βιομηχανικές δραστηριότητες. Ποια κενά μπορούμε να, να πληρώσουμε και τι είναι εκείνο που με τις πρωτοβουλίες μας μπορούμε να δραχθούμε ως ευκαιρία για να ενδυναμώσουμε το δυναμικό μας να πρικοδοτήσουμε το δυναμικό μας ώστε να προχωρήσουμε περισσότερο. Αυτά είναι πολύ πιο δύσκολα ερωτήματα να απαντηθούν είναι ερωτήματα τα οποία αναχώρα πρέπει να απαντηθούν, πιο εξειδικευμένα. Γι' αυτό είχαμε και την ε, ε, το γράφημα ή την εικόνα των νέων κινήτρων και των νέων συνόρων. Αλλά αυτά δείχνουν και σε σχέση και με την παλαιότερη τάση όσον αφορά τις ε, βιομηχανικές εξελίξεις, αυτοκινητόδρομους, σιδηρόδρομους, σε σχέση με την, ας το έννοια του ε, ανθρώπου που αγωνίζεται σε ένα μέτωπο New Frontiers, σε ένα νέο σύνορο το οποίο προσπαθεί να κατακτήσει. Ε, κατακτώντας ε, ε, χέρσες εκτάσεις τις οποίες καλλιεργούν και που μετά μπορούν να καταστήσουν παραγωγικές και που εμπεριέχουν δυνατότητες οικονομικής ανάπτυξης. Τηλεπικοινωνίες, το διαδίκτυο, αυτά είναι πράγματα τα οποία δεν υπήρχαν στο παρελθόν, δεν υπήρχαν ως κάτι το αυτονόητο. Από τις ε, τηλεπικοινωνίες ε, υπήρχε και άντληση κεφαλαίου, η δυνατότητα άντλησης κεφαλαίου για τις διάφορες συχνότητες, πράγμα το οποίο δεν υφίστατο παλαιότερα. Πρέπει να ε, υπάρξει η σωστή ρύθμιση, ένα σωστό ρυθμιστικό πλαίσιο εκμετάλλευσης συχνοτήτων για να μπορέσουν όλα αυτά να ανθίσουν. Και έτσι έχουμε εδώ, ας το πω έτσι, μία προσέγγιση ιδεατή ε, διανοητική θα έλεγα ώστε να μπορέσουμε να ενεργοποιηθούμε με τον καλύτερο τρόπο για να είμαστε παραγωγικοί. Να στρέψουμε το βλέμμα στο μέλλον, να δούμε ποιοι τομεί ε, θα πρέπει να αντιμετωπιστούν σε σχέση με την υγεία, την ε, περίθαλψη, την συνταξιοδότηση. Πώς ε, θα αντιμετωπιστούν όλα αυτά. Δεν έχω έτοιμε απαντήσει, αλλά αυτά είναι ερωτήματα τα οποία πρέπει να διατυπωθούν. Έχω μεγάλο κατάλογο εκείνων που ζητούν να παρέμουν. Θα διαβάσω τα ονόματα. Η ο συντάκτη νομοδότηση συντάκτρια και εκπρόσωπο των σοσιαλιστών και μετά όλος Λεσμίτα από του φιλελευθέρου και μετά έχουμε και ε, τον, συνάδελφο Χουντή από την Ενωτική Αριστερά και τον Χανς Peter Μάτιν από τους ε, μη εγγεγραμμένους. Θα ήθελα να είναι πιο σύντομοι τώρα οι συγητές στις απαντήσεις τους γιατί διαφορετικά δεν θα μπορέσουν να απαντηθούν όλα τα ερωτήματα. Απλά να επικεντρώνεστε στο, στον πυρήνα, στην ουσία του ερωτήματος και η ερώτηση πρέπει να απευθύνεται σε έναν μόνο από τους δύο εισηγητές μας γιατί διαφορετικά δεν θα τα καταφέρουμε. Υπερβάσουμε ρες, Παρακαλώ. Euh, Άκουσα αυτή την ε, έκκληση για το καπιταλιστικό σύστημα. Καταλαβαίνω την ε, λογική και το σκεπτικό. και δεν βλέπω να υπάρχουν ουσιαστικές ε, διαφορές. Αλλά υπάρχουν ορισμένα αντιφατικά στοιχεία. Δεν μπορούμε να λέμε από τη μία πλευρά ότι η κρίση είναι κρίση του τραπεζικού σήματος των G7 όπου η Ευρώπη είναι ο ουσιαστικός υπεύθυνος επειδή έχει αγοράσει προϊόντα χωρίς βάση τα οποία έχει παράγει το αμερικανικό δημοσιονομικό σύστημα. Είναι κάπως απλοϊκή η εξήγηση. Νομίζω ότι δεν είναι δυνατόν ε, να ακολουθήσει αυτή, αυτό το σκεπτικό κάποιος και να ξεχνά τελείως τις αμερικανικές ευθύνες. Δεν μπορούμε να είμαστε τυφλοί και να κοιτάμε απλούστατα τη μία απτυχή, του φακέλου που μας απασχολεί. Και συγχρόνως, και το γνωρίζετε πολύ καλά, εσείς οι ίδιοι λέτε ότι η πολιτική των αμερικανικών υποθηκών είχε ορισμένα μειονεκτήματα και ορισμένες αδυναμίες. Ουσιαστικά εγώ διαφωνώ άρδιν με τις δύο παρουσιάσεις που έγιναν διότι πιστεύω ότι υπάρχει ένα θέμα με το οποίο μπορώ να συμφωνήσω το ουσιαστικό γεγονός αυτής της κρίσης, το χαρακτηριστικό της, είναι ότι απέδειξε ε, σαν βασικό παίκτη στην αγορά τις ε, αναπτυσσόμενες χώρες, emerging countries, αναδυόμενες χώρες και το να πούμε ότι το θέμα είναι απλώς η καινοτομία δεν νομίζω ότι ε, κανένας διαφωνεί αλλά πέστε μου ποια μεγάλη επενδυτική τράπεζα προώθησε τους δύο αυτούς αναπτυξιακούς παράγοντες. Και έχω μία συγκεκριμένη ερώτηση για να επανέλθω στο θέμα του εργαστηρίου μας το οποίο είναι ότι μιλήσανε ε, κριτικά ε, επανειλημμένως και οι δύο μιλητές για τη Βασιλεία τι σας ενοχλεί στη Βασιλεία διότι ε, είπατε ότι θεωρείτε ότι η Ευρώπη πρέπει να τα βγάλει πέρα μόνη της δεν μπορούμε τίποτα να κάνουμε μαζί τουλάχιστον αυτό το μήνυμα εγώ αποκομίζω από τα σχόλιά σας θα παρακαλέσω και τον επόμενο να κάνει την ερώτησή του, Όλε Σμιτ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για τις παρεμβάσεις. Ε, παρόλο που είναι κάπως ε, απεσιόδοξες και μας, διαγράφουν, μας περιγράφουν μία πολύ μαύρη και σκοτεινή εικόνα. Δηλαδή ότι μας περιμένουν ακόμη χρόνια ε, με τέτοια ατυχή γεγονότα και πρέπει να σας πω ότι ο κόσμος είναι καλύτερος από όταν, όταν ήμουν εγώ 20 ετών υπάρχει περισσότερη ελευθερία πιστεύω ότι η παγκοσμιοποίηση έχει κάνει και καλά και αυτό είναι κάτι που πρέπει να λεχθεί ένα βασικό μου ερώτημα είναι ότι είπατε ότι ο Κέινς έχει πεθάνει κάποια στιγμή όλοι θα πεθάνουμε ε, τέλος πάντων γιατί οι αγορές δεν κατάφεραν να αυτορυθμιστούν και να αυτοδιορθωθούν εάν υπάρχει πραγματικός καπιταλισμός και ελεύθερη αγορά ε, διότι ε, ορισμένοι είναι πολύ απογοητευμένοι με τις επιδόσεις τους. Οπότε ε, θα ήθελα να μου πείτε τι γίνεται και το άλλο μου ερώτημα δεν αναφέρεται εις ε, τις Ηνωμένε Πολιτείες αλλά βλέπω ότι οι Ηνωμένε Πολιτείες είναι τώρα στενά συνδεδεμένες με την Κίνα και όλοι έχουμε στενούς συσχετισμούς. Αν υπάρχουν λοιπόν 500 εκατομμύρια Κινέζοι που ζουν με 2,5 δολάρια την ημέρα και άλλα 800 ε, ε, εκατομμύρια ζουν με 1,5 δολάριο την ημέρα και έχουν 4 εκατομμύρια οι Κινέζοι σημαίνει ότι υπάρχει μια τεράστια αγορά και τώρα φτάνω στην συγκεκριμένη ερώτηση που μου ζητά ο πρόεδρος. Δηλαδή, τι μπορεί να κερδίσει και η Ευρώπη από αυτήν την τεράστια αγορά. Δηλαδή, να βγάλει κάτι και η Ευρώπη και όχι μόνο οι Ηνωμένε Πολιτείε. Νομίζω ότι αν είμαι σύντομος θα είμαι πιο ορθολογιστικός από ό,τι συνήθως. Όταν είπα ότι η κρίση αυτή χρειαζόταν, Ίσως θα μπορούσαμε να είχαμε αποφύγει μία μεγαλύτερη κρίση αν είχαμε δεχθεί νωρίτερα μικρότερες κρίσεις. Ο Γκρίσμαν είναι απογοητευμένος και αντιλαμβάνομαι γιατί, διότι όποτε υπήρξε μία ύφεση στην Αμερικανική οικονομία στο δεύτερο ήμιση της δεκαετίας του 90 και στην αρχή της δεκαετίας του 2000 έριχναν στην αγορά ε, χρήματα με χαμηλά επιτόκια. Για να αποφύγουμε λοιπόν τις μικρές κρίσεις ε, οικοδομήσαμε ε, δάνεια τα οποία οδήγησαν σε μια μεγάλη κρίση και ε, πρέπει να δεχθούμε σε αυτή την οικονομία αγορά, στο σύστημα αυτό το καπιταλιστικό, ονομάστε το όπως θέλετε, ότι πρέπει να δεχθούμε μικρότερες κρίσεις για να αποφύγουμε μία μεγαλύτερη. Δηλαδή βρισκόμαστε σε μια αυστριακή κατάσταση. Νομίζω ότι αυτή είναι η καλύτερη ε, εξήγηση. Δεν έχει καμία σχέση ε, με την τωρινή Αυστρία αλλά ο Αυστριακός πέτερ, είχε πει ότι αν υπάρχει υπερβολική επένδυση, χαμηλά επιτόκια και μεγάλη ρευστότητα στην αγορά υπάρχει κρίση, οδηγεί σε κρίση. Έχουμε λοιπόν δημιουργήσει ένα πλεονεσμα κατασκευαστικό στην, ε, σε ολόκληρο τον κόσμο τα τελευταία 20 χρόνια και το έχω πει στην χαλιβουργία, διότι ε, από το τέλος του Σοβιετικού Μπλοκ μέχρι το 2000 το ΚΑΠΕΞ, δηλαδή οι κεφαλαιοχικές δαπάνες τριπλασιάστηκαν δηλαδή ε, δημιουργήσαμε ε, μία ε, ένα πλεόνασμα 15% εάν θεωρήσουμε ότι στο παρελθόν καλύπταμε τη χρήση του 100% της παραγωγής πράγμα το οποίο δεν συνέβαινε και ε, ε, ε, γι' αυτό υπάρχει και το θέμα του πληθωρισμού για τα επόμενα χρόνια. Τώρα, όσον αφορά την ε, πολιτική ε, κόστους ε, των κατοικιών. Οι Αμερικανοί βοηθώντας την τράπεζα δεν ήθελαν να, χρηματοδοτήσουν την κρίση. Οι δύο οργανισμοί δανειοδοτικοί οι οποίοι παρέμειναν αποφάσισαν να παραμείνουν σαν μία τράπεζα και θα δούμε πού θα πάνε. Όσον αφορά τη Βασιλεία που ζητά μεγάλο ποσοστό ενεργητικού προς το δάνειο, εγώ συμφωνώ να υπάρχει υψηλό ποσοστό ε, μεν και πιστεύω ότι το σύστημα λειτουργεί καλά και πρέπει να το δεχτούμε. Δεν μου αρέσει η στάση που έχουν ορισμένοι στις Βρυξέλλες και σε ορισμένες εθνικές κυβερνήσεις που αντιτίθενται διότι ξέρουν ότι ε, δεν υπάρχει δυνατότητα για ορισμένες ε, τράπεζες να καλύψουν τις ε, εγγυήσεις για τα δάνεια που θέλουν βάσει αυτών των ποσοστών. Ε, πιστεύω ότι ακόμη ε, υπάρχει ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι που ζουν με δύο δολάρια την ημέρα αλλά όχι πλέον στην ε, Κίνα και όσον αφορά τα αποθέματα της ε, Κίνας τα 4-3 τρισεκατομμύρια εκ των οποίων ένα μεγάλο ποσοστό είναι σε δολάρια και θα παραμείνει για τα επόμενα έτη εάν δεν βρεθεί εναλλακτικό αποθεματικό νόμισμα ε, ε, λέτε γιατί δεν μπορεί να αναβαθμιστεί η Ευρώπη. Ε, για τους πρώτους μήνες ε, οι εξαγωγές της ε, Γερμανίας προς την Κίνα ήταν μεγαλύτερες από τις εξαγωγές της Γερμανίας στην Γαλλία. Δηλαδή πολλές ευρωπαϊκές χώρες εποφελούνται από το τι γίνεται στην Κίνα και θα μπορέσουμε έτσι να βοηθηθούμε να βγούμε από την κρίση μέσω αυτών των αναδειωμένων αγορών. Ο κύριος Μέισον ε, όσον αφορά το ρόλο των ε, ε, επενδυτικών τραπεζών ε, σε σχέση με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ούτω καθεξής. Όσον αφορά τη Βασιλεία, ένα βασικό θέμα είναι ότι είναι περισσότερο κρίσης χρεών παρά ενεργητικού. Δηλαδή υπήρχε πάντοτε χρηματοδότηση των δημοσιονομικών οργανισμών και συμφωνώ με τον προλαλήσαντα ότι υπήρχαν πάντοτε κρίσεις ε, στα τελευταία 15 χρόνια είχαμε 8 έως 10 κρίσεις ε, τις οποίες όμως θεωρούσαμε υποσιώδεις και γι' αυτό ε, τις παραβλέψαμε μέχρι ότου φτάσαμε σε ένα σημείο τόσο μεγάλης κρίσης. Και όσον αφορά την αναθεώρηση της Συμφωνίας της Βασιλείας ε, πρέπει να παρακολουθεί τα εχέγγυα μεν της χρηματοδότησης αλλά ε, πρέπει να δούμε ε, ε, πώς πρέπει κανείς να εξετάζει την πιστοπληστική αξιολόγηση για κάποιο ομόλογο και ούτω καθεξής και επίσης την μόχλευση πορών τραπεζικών ε, ιδρυμάτων διότι υπάρχουν ε, διάφοροι τομείς ε, οι οποίοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν εχέγγυα για να διευρύνουμε τα δάνεια διότι ε, πρέπει να βοηθήσουμε τις τράπεζες να συνεχίσουν να δανείζουν. Άρα πρέπει να ε, εξασφαλίσουμε ότι θα δημιουργούμε ε, νέα εχέγγυα, νέες εγγυήσεις και ότι θα εξυπηρετούμε τις υπάρχουσες εγγυήσεις και υποθήκες. Επίσης πρέπει να δούμε τον ρόλο των επενδυτικών τραπεζών και της Κίνας όπως είπατε. Ε, νομίζω ότι οι τράπεζες εποφελούνται από την ανάκαμψη της αγοράς. Πολλές τράπεζες δεν χρειάστηκαν βοήθεια διότι εμείς ε, δώσαμε βοήθεια στην Αμερική η οποία ήταν εισάξια με αυτήν πριν τη του 1929 χωρίς να έχουμε φτάσει στο ίδιο σημείο. Και όσον αφορά την Κίνα, η Κίνα φροντίζει για την Κίνα και κανείς άλλος. Αν πήγατε στην Αφρική, αν κοιτάξετε γύρω στην Αφρική, βλέπετε ότι στην εξορρυκτική βιομηχανία χρησιμοποιείται ε, ε, εξοπλισμός κινέζικος, προσωπικό κινέζικο και δεν δίνουν τίποτα στην Αφρική. Ε, θα μιλήσω περισσότερο για το ε, χρέος και το το μετοχικό κεφάλαιο και την εξίσωση αυτών δύο. Ε, το φορολογικό σύστημα ε, θα πρέπει να αλλάξει στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες ε, Πολιτείες. Επίσης μιλήσατε για το κεφάλαιο κινδύνου. Στην ε, Ευρώπη βασιζόμαστε πάρα πολύ στο χρέος για να χρηματοδοτήσουμε τις νέες επιχειρήσεις. Ε, γιατί έχουν ε, πρόβλημα οι επιχειρήσεις αυτές να έχουν πρόσβαση σε μετοχικό κεφάλαιο. Έχετε άποψη επίσης και για την οδηγία για τα hedge funds θα έχει αρνητικές επιπτώσεις για το κεφάλαιο κινδύνου. Και πώς μπορούμε εμείς να προωθήσουμε το κεφάλαιο κινδύνου στην ευρωπαϊκή υπηρεσία της Ευρωπαϊκής ευρωπαϊκές Πράγματι, οι δύο εισηγήσει ήταν ενδιαφέρουσες. Πριν κάνω όμως τη συγκεκριμένη ερώτηση που, με ρωτήσατε, που είπατε για να συντομεύσουμε τον χρόνο, θέλω να σας κάνω μια εξομολόγηση. Αυτό που διέκρινα και από τις δύο εισηγήσει είναι μια απέραντη βεβαιότητα και σιγουριά για τα συμπεράσματα που έχουν εξαχθεί και για το τι πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα. Δεν ξέρω πώς επηρεάζουν τις σκέψεις των κυβερνήσεων, των κυβερνώντων στις ΗΠΑ. Πολιτείες. Αλλά θα ήθελα να ρωτήσω και τους δύο, ιδιαίτερα τον δεύτερο, τον κύριο Γιούκεν. Μετά την κρίση, δεν αμφιβάλλει καθόλου ότι αυτά που λέει ίσως οδήγησαν στην κρίση. Δεν τα βάζει καθόλου στην κριτική αν πράγματι είναι σωστά, γιατί κατά τη γνώμη μου όλα αυτά που λέει ήταν που οδήγησαν στην κρίση. Αλλά αυτή είναι μια αξιολόγηση. Δεν βλέπω να βγαίνουν τα συμπεράσματα. Με παραξένεψε η βεβαιότητα και ήθελα να σα το ξεμολογηθώ. Το δεύτερο το συγκεκριμένο ερώτημα που θέλω να κάνω είναι πώ αξιολογούν και οι δύο εισηγητέ τη συμμετοχή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στο μηχανισμό στήριξη χωρών που έχουν προβλήματα στην Ευρωζώνη είναι μορφή διατλαντικής συνεργασίας για το ξεπέρασμα της κρίσης. Και η επιμέρους ερώτηση είναι η εξής. Αν άκουσα καλά τον κύριο Γιούγκεν, είπε η Ελλάδα ποτέ με όλα αυτά που κάνει δεν θα ξεπληρώσει το χρέος. Τότε, η... τότε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο τι κάνει κύριε, ρισκάρει τα χρήματά του που δεν θα πάρει ποτέ. Σας ευχαριστώ. Για την πρώτη ερώτηση. Έχετε απόλυτο δίκιο όσον αφορά το καθεστώς, ε, όσον αφορά την ε, φορολογία και το φορολογικό βάρος. Έχουμε συνεισφέρει στην κρίση. Είμαστε υπέρ ενός ε, φορολογικού καθεστώτος που είναι υπέρ της χρέωσης, ευνοεί την υπερχρέωση και το ίδιο ισχύει και σε σχέση με την πολιτική ε, για τα φορολογικά θέματα. Ο κύριος λόγος, επειδή το, το κεφάλαιο κινδύνου, ας το πω έτσι, είναι υπανάπτυκτο ακόμα, κατεφημισμών κιόλα στην Ευρώπη. Αυτό είναι ένας λόγος. Πρέπει λοιπόν να φύγουμε από την ε, αρνητική αντιμετώπιση ε, φορολογικά και να μην ευνοούμε την υπερχρέωση. Το αντίθετο πρέπει να κάνουμε. Και όσον αφορά την ε, ε, υπανάπτυξη όσον αφορά το 35 έως 38 35 έως 38 ε, τρισεκατομμύρια κεφάλαια κινδύνου όσον αφορά που ε, στην Ευρώπη είναι 3,4 έως 4, 3,4 έως 4 σε σχέση με τις ΙΠΑ. Ε, Αν δει κανεί αυτή την αναλογία, 1 προς 10 ή 10 προς 1 είναι δυσανάλογη. Έχουμε λοιπόν απουσία καινοτομίας στις επενδύσεις και δόξα τω Θεώ οι επενδυτικές τράπεζες δεν είχαν ε, ε, εμπλακεί όσον αφορά την χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Θα είχαμε τεράστια προβλήματα. Δεν τις χρειαζόμαστε γι' αυτό. Χρειαζόμαστε την ε, μεταλαμπάδευση του πνεύματος του επιχειρήν όσον αφορά τους αγγέλους του πνεύματος του επιχειρήν. Και φυσικά η κατάσταση αυτή στο, στην οποία έχει καταλήξει η Ευρώπη και για την προσπάθεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να συνεισφέρει στην αντιμετώπιση του προβλήματος. Ένα στοιχείο, η ιδέα να υπάρξει ένα σύστημα επιτήρησης και όσον αφορά τις επενδυτικές προσπάθειες και το κεφάλαιο κινδύνου όταν θα απασχολούν 50 ή παραπάνω απασχολούμενους. Κανένας δεν θα έπαιρνε τα χρήματα από αυτούς γιατί δεν θέλει κανείς να εμπλέκεται σε μια τέτοια διαδικασία ε, ενημέρωσης όσον αφορά τους ανταγωνιστές και το πού βρίσκεται μια επιχείρηση σε σχέση με τους ε, ανταγωνιστές της. Αν ε, κάτι τέτοιο συμβεί, τότε θα θανατωθούν οι προσπάθειες καινοτομίας και θα ενθαρρυνθούν άλλοι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης να ξεκινήσουν εκείνοι κάτι. Και για την ανάπτυξη σε νέων επιχειρήσεων για την ε, Angel Investment θα βλέπαμε πολύ λιγότερες επιχειρήσεις να ξεκινούν. Αν θέλετε με αυτόν τον τρόπο αυτή ε, τη ρυθμιστική προσπάθεια να ξεκινήσετε ε, θα έχετε λιγότερες ε, επιχειρήσεις που θα ε, ξεκινούν τις δραστηριότητές τους και αυτό θα ήταν η τορπίλη που θα τορπίλιζε τις επενδυτικές προσπάθειες στην Ευρώπη. Είμαστε ήδη υπανάπτυκτοι σε σχέση με αυτό και ποιος θα ήθελε να υπονομεύσει ακόμα περαιτέρω. Ελπίζω ότι απάντησα όλες σας τα ερωτήματα. Ευχαριστώ. I didn't answer this one. Yes, was on... Το απάντησα αυτό. Έχετε δίκιο. Είμαι στην επόμενη σελίδα. Σωστό. Σε σχέση με τα αίτια για την κρίση, δεν είμαι βέβαιος αν κάνατε λόγο για τις ε, δυσαναλογίες ε, οι μη ισόρροπες σχέσεις στην Ευρώπη ή την κρατική υπερχρέωση ή αν αναφέρεστε στην κρίση των χρηματοπιστωτικών, χρηματοοικονομικών αγορών. Ε, αυτή τη χρονική στιγμή δεν ξέρει κανείς ακριβώς σε τι αναφέρεται κάποιος όταν αναφέρεται στην κρίση. Αλλά εδώ πρέπει να δούμε το θέμα των απαντήσεων για το 75% ε, στην Ευρωζώνη, 105% σε σχέση ε, με την λέσχη των 7% και θα η Ιαπωνία είναι πάνω από το 200 και το Ηνωμένο Βασίλειο πάει στο 107 όσον αφορά την υπερχρέωση. Και υπάρχουν και αίτια τα οποία έχουν οδηγήσει σε αυτή την κρίση και σε αυτή την ε, αναταραχή. Τις προάλλες είχαμε μια ε, διάσκεψη και είχαμε και τον κύριο οικονομολόγο της Goldman Sachs. Τα καλά μαντάτα είναι, τα, τα, τα κακά νέα είναι κακά για την Ευρώπη. Τα καλά νέα είναι ότι δεν έχει επίπτωση αυτό στην ε, παγκόσμια οικονομία, μια και η εμβέλεια αυτού, αυτής της συνιστώσας είναι μικρή γνωρίζετε ότι ήμουν ο πρώτος στις Βρυξέλλες που είχε προτείνει να έχουμε ένα ευρωπαϊκό νομισματικό ταμείο που θα δρά όχι όμως για να διασώζει χώρες αλλά προληπτικά να δρά. Χρειαζόμαστε λοιπόν ένα καθεστώς για η αλληλεγγύη είναι αμφίδρομος δρόμος, δεν είναι μονόδρομος. Τώρα αν τον Διεθνές Νομισματικό Ταμείο θα κάνει όλη τη δουλειά, θα φτάσει μέχρι τέλους δεν το γνωρίζω. Το πιο σημαντικό όμως στοιχείο είναι όχι αυτό το οποίο εγώ έχω υπόψη μου το τι θα κάνει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Είναι το πιο σημαντικό να μπορέσει να υλοποιήσει η Ελλάδα τις υποχρεώσεις της και να έρθει στο ύψος των περιστάσεων σε σχέση με τις υποσχέσεις που έχει αναλάβει η ελληνική κυβέρνηση. Αυτό είναι στοιχείο που έχει σημασία κλειδιού. Αν η Ελλάδα το 2013 ή το 2014 καταλήξει με 145 ή 150 ε, ε, ε, αναλογία χρέους όσον αφορά το ΑΕΠ, βλέπουμε ότι εδώ υπάρχει περίοδος χαμηλών επιτοκίων Τέλειωσε τώρα αυτό, υπάρχει υψηλότερο επιτόκιο για η μεγαλύτερη χρέωση και το ίδιο θα ισχύσει και για φέτος και του χρόνου και για το 2011. Και το ΑΕΠ θα συρρυκνώνεται. Και τι θα γίνει. Θα έχουμε μια κατάσταση όπου ουσιαστικά θα βλέπουμε ότι ο, ο, νομαστής και ο παρανομαστής θα αλλάζουν ε, ε συσχετισμό ή αναλογία. Θα υπάρχει για παράδειγμα συρρύκνωση και τότε θα ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα. Εγώ θα έλεγα είναι προς το καλύτερο συμφέρον της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης να χρησιμοποιηθεί ο χρόνος που εξαγοράζεται τώρα για να επιτευχθεί μια αναδιάρθρωση, μια αναδιάρθρωση μέσα σε σωστά πλαίσια και με σωστές, ε, σωστούς στόχους. Και έτσι λοιπόν θα έλεγα η ε, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα μπορέσει να συνεισφέρει. Πιστεύω ότι αυτό είναι και μια ένδειξη το ότι στοχεύουμε σε μια βελτίωση της κατάστασης. Ευχαριστώ. Θα απαντήσω τις ερωτήσεις αυτές με την αντίστροφη σειρά όσον αφορά την αισιοδοξία που φαίνεται να εκπλήσει. Ναι, η αισιοδοξία είναι κάτι το θα έλεγε κανείς στρεβλό. Όμως παρόλα αυτά τι βλέπουμε. Βλέπουμε ότι ε, υπάρχει αυτή η τάση, βλέπουμε παραγωγικότητα να αυξάνεται εργάζονται σκληρότερα οι εργαζόμενοι για να διασφαλίσουν και να κρατήσουν τις θέσεις απασχόλησής τους. Το σύστημα λοιπόν λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο, έστω και αν αυτό δεν είναι κάτι το οποίο ευχαριστεί τους πάντες. Λειτουργεί λοιπόν το σύστημα και η ε, αποκάλυψη στοιχείων όσον αφορά τις ε, ε, τιμές είναι ίσως ένα στοιχείο το οποίο κάποιους ανησυχεί. Εκείνο το οποίο πρέπει να δούμε είναι η δημογραφική φούσκα. Έχουμε μεγάλη εξάρτηση σε σχέση με το συνταξιοδοτικό μας σύστημα για από ένα συρρυκνούμενο αριθμό εργαζομένων. Και έχουμε εδώ και spreads τα οποία οδήγησαν συνταξιοδοτικά ταμεία και ε, θεσμικούς επενδυτές να οδηγηθούν σε ε, δημιουργία φούσκας και ε, δυσανάλογες ε, καταστάσεις. Είναι εδώ ένα θέμα ζήτησης θεσμικών επενδυτών όταν βλέπουμε ότι οι θεσμικοί επενδυτές ε, ε, θέλουν να πετύχουν μεγαλύτερη κερδοφορία από ό,τι σε σχέση με τα κεφάλαια τα οποία έχουν συγκεντρώσει. Και βλέπουμε εδώ ότι δημιουργούν έτσι με αυτόν τον τρόπο φούσκες. Όσον αφορά όμως την ανάπτυξη, ποιος είναι εκείνος ο οποίος ε, αγοράζει το χρέος. Είναι ένα ερώτημα που πρέπει να δώσουμε προσοχή στην ε, αναθεώρηση της Συμφωνίας Βασιλείας ε, στην τρίτη φάση. Να δούμε τι γίνεται σε σχέση με τα θεσμικά αποθέματα και τους θεσμικούς επενδυτές. Το Bureau of Indian Affairs για παράδειγμα στις ΕΠΑ και την ε, κακοδιαχείριση των ε, κεφαλαίων που τους είχαν ε, χρησιμοποιούσαν ως διαπίστευμα για τους ε, ε, ηθαγενείς Αμερικανούς, ε, τους ερυθρόδερμους. Και με αυτόν τον τρόπο λοιπόν η εγγύηση της Αμερικανικής κυβέρνησης, ακόμα και αν η Αμερικανική κυβέρνηση εμπλέκεται, το πρόβλημα παραμένει. Το θέμα είναι τι γίνεται σε σχέση με, τις, με τα κεφάλαια για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Είναι κάτι ε, όσον αφορά την ε, τελευταία νομοθεσία ε, της, ε, στις για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, το νομοθετικό πλαίσιο για την ε, δημιουργία ενός πλαισίου υποστήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που εγκαταλείφθηκε εντωμεταξύ όμως τα βαρύδια αυτά βάριναν την Αμερικανική οικονομία. Μια καλύτερη ίσως προσέγγιση είναι να διασφαλίζεται αυτή η διαφάνεια όσον αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις όπως και στις ΗΠΑ, δίνοντας έναν πίνακα ή ε, έναν ε, κατάλογο ε, επιδόσεων των μικρών επιχειρήσεων. Είναι μια κατεύθυνση που χρησιμοποιήθηκε και από την Αργεντινή και από ό,τι φαίνεται έχουν επιτευχθεί αποτελέσματα θετικά. Τελευταίοι δύο αγορητές, Χάς Πέτερ Μάρτιν και Ρόνατα Χίμνερ. Ευχαριστώ. Στην παρουσίασή σας είχατε πει ότι κάθε, χώρα έχει, πρέπει να χρησιμοποιήσει τους δικούς της πόρου και δεν υπάρχει μια συνταγμή για όλους. Ε, θα πρέπει να το κάνει ο καθένα μόνο του ή να αναγκαστεί να το κάνει, α πούμε, παραδείγματο χάρη μέσω ενό παγκοσμίου πολέμου. Μπορείτε να μα το εξηγήσετε, ε, Μπορείτε να μα το εξηγήσετε λιγάκι αυτό. Ε, τι ρόλο θα μπορούσε να παίξει η Ευρώπη εκεί και τι εννοείται με αυτό το παγκόσμιο πόλεμο. Κύριε Γιούγκεν, υπάρχουν πολλά σημεία που μπορούμε να συμφωνήσουμε. Με αυτή την ανάγκη να ανοίξουν πολλές ευρωπαϊκές χώρες στην επιχειρηματικότητα. Αν το κάνουμε αυτό, είπατε ότι θα πρέπει να έχουμε 5 εκατομμύρια επιπλέον επιχειρηματίες. Παρ' όλα αυτά θα έχουμε πολλούς ανθρώπους που δεν θα μπορέσουν να βγάλουν τα προς το ζήν με τα συνήθη μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας τώρα. Η ιδέα σας ή η συνταγή σας δεν λέει ότι θα πρέπει να εγκαταλείψουμε το γερμανικό μοντέλο και να ακολουθήσουμε το βιετναμέζικο μοντέλο. Και αν ναι, τι σημαίνει αυτό για την πολιτική κουλτούρα που έχουμε στην Ευρώπη. Όλα τα πολιτικά κόμματα, με ελάχιστε εξαιρέσει, δεν ψηφίστηκαν για να πάνε στην εξουσία υποσχόμενα το αντίθετο από αυτό που λέτε εσείς. Άρα δεν θα πρέπει να αμφισβητηθεί όλο το πολιτικό ε, και κομματικό σύστημα. Έπειτα υπάρχουν πολλές αναφορές για σπέκουλα εναντίον του, ευρώ, του ευρώ. Κακή σπέκουλα. Ποιο είναι το ποσοστό της κακής σπέκουλας ε, κατά την εκτίμησή σας. Και πέστε μας, ε, ποιο είναι το κακό στοιχείο της σπέκουλας εναντίον του ευρώ. ξέρουν όλοι τι εννοείται με αυτό το βιετναμέζικο μοντέλο. Εννοείται μήπω την Κορέα. Όχι, είναι πιο προχωρημένοι οι Βιετναμέζοι. Υπάρχουν περισσότεροι νέοι, α πούμε. Ε, θέλουν να κάνουν επιχειρήσει. ε, κάνουν, προσπαθούν να κάνουν τα πάντα για να βγάλουν λεφτά οι Βιετναμέζοι. Νέοι, ε, ρίχνονται σε νέε επιχειρήσει κτλ. Προ τον κύριο Χιούγκεν. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να βγει κανεί από μια κρίση. Μάλλον θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι αυτό που κάναμε στην Ευρώπη είναι ότι επιλέξαμε το μονοπάτι της περισσότερης, των περισσότερων κανόνων και ρυθμίσεων για να διορθώσουμε τις αποτυχίες των αγορών και α, των κυβερνήσεων. Έπειτα, η διάστησή σας, τι σας λέει. Θα τα καταφέρουμε με αυτό το μονοπάτι που ακολουθούμε με τους περισσότερους κανόνες. Ή θα δημιουργήσουμε ένα σύστημα που θα είναι πιο ευεπίφορο σε κρίση. Επίσης, δεν αντιλαμβανόμαστε την περιπλοκότητα, την περίπλοκη φύση από ό,τι φαίνεται του χρηματοπιστωτικού τομέα και ούτε της, του τρόπου διαχείρισης των ε, επιχειρήσεων. Προς τον κύριο Μέισον. Όταν μιλάτε για το μεγάλο κόστος ε, που θα πληρώσουμε αν ε, κάνουμε κάτι λάθος τώρα, Μιλήσατε για αυτή την, το δίπολο, ας πούμε, αφαιρεγκαιότητας και έλλειψης ρευστότητας. Μπορείτε να δώσετε περισσότερες εξηγήσεις. Παρακαλώ, τρία λεπτά το πολύ στις απαντήσεις σας. Νομίζω ότι αυτό είναι πολύ ώρα. Τώρα κατάλαβα τι εννοείτε μιλώντας για τους Βιετναμέζους. Δεν ξέρω ποιο είναι το γερμανικό πρότυπο για να είμαι Ενδεχομένως υπάρχουν διάφορες ερμηνείες και ο καθένας τις χρησιμοποιεί. Είναι σαν το ευρωπαϊκό κοινωνικό πρότυπο και ε, πιστεύω ότι το ευρωπαϊκό κοινωνικό πρότυπο δεν είναι ευρωπαϊκό γιατί έχετε πολλά κρατημέλη, δεν είναι κοινωνικό και δεν είναι πρότυπο για κανέναν. Όσον αφορά τώρα τους Βιετναμέζουν, οι Γερμανοί πρέπει να είναι πιο επιχειρηματικοί, ε, θα πρέπει έχουν μία μείωση εκινήσεως επιχειρήσεων. Πέρυσι ήταν το πιο χαμηλό σημείο από το 1995 και όσον αφορά τους κύκλους και αν υπάρχει μία συνέπεια και συνέχεια όλοι μπορεί να φτωχύνουμε αλλά αν το γνωρίζουμε ε, χρειαζόμαστε περισσότερη καινοτομία και χρειαζόμαστε τους επιχειρηματίες για να προσφέρουν δυναμικά δυναμισμό για να υπάρξει ε, ένταξη ε, περισσότερων ε, ανθρώπων στη διαδικασία και λιγότερης πατάλης χρημάτων. Μετά, αναφερθήκατε στην κερδοσκοπία κατά του ευρώ. Δεν ξέρω τι θα πει speculation, θα πει ουσιαστικά ανάλυση της καταστάσεως και ε, ε, όσοι, πουλούν ε, short κάτι είναι καλύτεροι από τις, τους οίκους πιστοληπτικής αξιολόγησης. Πάρτε τη Lehman Brothers, όλοι πουλούσαν τις συμμετοχές της, οπότε δεν χρειαζόταν κανείς rating agencies, οπότε... Αντιλαμβάνεστε τι γίνεται όταν ξεπουλάει κανείς, πράγμα το οποίο βέβαια είναι πάρα πολύ επικίνδυνο διότι εάν προπολεί κανείς short πρέπει κάποια στιγμή να ξαναγοράσει και βλέπω ότι αυτή τη στιγμή σε υψηλό επίπεδο γίνεται συζήτηση για γυμνό short, ντυμένο short. Δεν θέλω να ακολουθήσω αυτές τις συλλογικές αλλά αυτό που έχω να σας πω είναι χωρίς να αυξήσω τους φίλους μου λέγοντας αυτά, ε, ίσως επαναλαμβάνω κάτι που έχει ήδη λεχθεί. Οι short sellers και οι καιροσκόποι έχουν επιτύχει περισσότερα στις τελευταίες 12 εβδομάδες από η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα, ε, οι Υπουργοί του ΕΚΟΦΗΝ σε 12 χρόνια όσον αφορά το δημοσιονομικό καθεστώς, τη συζήτηση για το δημόσια χρέη ε, και ε, χάρη εις τους καιροσκόπους επιτεύχθηκαν όλα αυτά. Άρα δεν θέλω να ε, διαχωρίσω τους κακούς καιροσκόπους από τους καλούς, απλούστατα να διαχωρίσω μεταξύ τους των πιο επιτυχών και των λιγότερο επιτυχών. Διότι ορισμένοι ουσιαστικά υπάρχουν χάρη στα ευρωπαϊκά προγράμματα. Αγόρασαν ομαδικά ομόλογα και είχαν υψηλότερα επιτόκια από ό,τι στα γερμανικά Bund και μετά από 5-8 χρόνια σωστά υπολόγισαν ότι δεν θα τους εγκατέλειπαν οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και άρα όντως ε, πρέπει να δούμε εάν πρέπει να επιτρέπουμε αυτές τις συλλογιστικές. Κυρία Χίμπνερ, ε, το αν χρειάζεται περισσότερη νομοθεσία, αν ε, υπάρχει σχέση μεταξύ δυναμικής ανάπτυξης και νομοθεσίας είναι κάτι που πρέπει να συζητήσουμε, αλλά η ιστορία δεν επαναλαμβάνεται, διδάσκει όμως. Και αυτό το οποίο μας διδάσκει είναι ότι ακόμη και αν κάποιος δεν θέλει να διδαχθεί, βλέπουμε ότι πάντοτε μετά από μία κρίση υπάρχει χαμηλό επίπεδο ανάπτυξης λόγω της πιο αυστηρής νομοθεσίας. Και μετά από μερικά χρόνια λένε ορισμένοι, ε, μπορούμε να τα καταργήσουμε αυτά και αρχίζει και πάλι η κατάσταση να δείχνει καλή, υπάρχει μία υπερεκτίμηση του κινδύνου, υπερεκτίμηση των ικανοτήτων κάποιου να βρει το σωστό σημείο να επενδύσει, ε, υπερβολική χωρητικότης επένδυση, ε, μία καλοπροαίρετη οικονομία όπως στην εποχή του Greenspan, αυτός είναι ο κύκλος και έχει λεχθεί ότι ο επόμενος κύκλος θα είναι το 2018. Γιατί? Γιατί τότε αυτοί που είναι υπεύθυνοι σήμερα είτε έχουν ξεχάσει, είτε είναι άνεργοι, είτε δεν γνωρίζουν ποια, είναι, ποια ήταν η κρίση και ε, γι' αυτό μπορώ να σας πω ότι τα πράγματα δεν αλλάζουν τα τελευταία 800 χρόνια οι κρίσεις είχαν τα ίδια χαρακτηριστικά. Το, τα γράφονται αυτά σε ένα βιβλίο που πολύ μ' αρέσει. Είτε μιλάμε για το Μισισιπί, είτε για οτιδήποτε. Το 1887, το 1900 κάτι, κάθε μερικά χρόνια όταν οι επόμενοι ευρωβουλευτές θα είναι εδώ θα ακούσουν πάλι μία δόση από τα ίδια. Μην ανησυχείτε. Ευχαριστώ. Ε, αν θέλετε να πάτε λίγο πιο πίσω στην ιστορία όσον αφορά την ερώτηση που τέθηκε εις ε, τον Warren Neal ε, στο London School of Economics βλέπουμε ότι κανείς γίνεται πολύ δημιουργικό σε εποχή πολέμου και αυτό απέδειξε η παγκόσμια ιστορία. Υπάρχει και ένα βιβλίο του Freeman and Schwartz σχετικά με την την παρακολούθηση ε, της ε, ε, οικονομίας στην Αμερική όπου βλέπουμε ότι οι καταστάσεις επαναλαμβάνονται και ε, πρέπει κανείς να εξετάσει την αλληλοσχέτιση ε, της οικονομικής και της κοινωνικής πτυχής διότι ε, αυτό το οποίο διαπιστώνουμε τώρα είναι οι κοινωνικές πτυχές δηλαδή πολίτες που δεν μπορούν να ανταποκριθούν και προσπαθούν να επιτύχουν αλλά με μεγαλύτερο κοινωνικό κόστος και τέλος πρέπει να δούμε ε, ποιο είναι το ε, επίπεδο της ανάπτυξης που θα, ε, θα επιτύχει η ζεύξη. Διότι ίσως θα μπορέσουμε να συνδυάσουμε προχωρήσουμε με διαφορετικά μέτρα και σταθμά για τις ε, αναπτυσσόμενες χώρες, για τις χώρες μικρής αναπτύξεως και τις ε, BRICS. Λοιπόν, έχει, έχει κανείς ε, εξετάσει την ε, ανάλυση της παγκοσμίου οικονομίας κατά την ε, εποχή του, της κρίσης του 1929 όπου είδαμε ότι οι τράπεζες δεν απέτυχαν και δεν χρεοκόψαν από τόμος από τη μια μέρα στην άλλη αλλά επί εβδομάδες για να μην σας πω επί χρόνια πριν έστελναν οι νομοθέτες ε, γράμματα, έβαζαν πινακίδες, ζητούσαν από τις τράπεζες να μειώσουν τους κινδύνους που ανελάμβαναν. Άρα ποιοι απέτυχαν οι τράπεζες αυτές. Οι άλλες οι τράπεζες οι οποίες ε, ήταν πιο σόφρονες δεν απέτυχαν η κρίση ρευστότητος ε, στην ελληνική οικονομία ουσιαστικά κράτησε δύο ημέρες. Αλλά αυτό δεν ισχύει ε, και μπορείτε να μου το αποδείξετε διότι ε, εγώ αν μου αποδείξετε ότι δεν έχω δίκιο θα κερδίσω. Δεν είτε πρόκειται για την κρίση ρευστότητος ή στην εποχή του 1929 βλέπουμε ότι όντως και εκεί υπήρχε ε, κρίση οξία για δύο μέρες. Αλλά Τώρα, εάν κάποιος είναι αφερέγγιος δεν θα τον ε, βοηθήσει καμία τράπεζα. Οπότε εμείς αυτό που ζητάμε από τους νομοθέτες είναι να προλάβουν πριν φτάσει η τράπεζα να μην δανείζει πια. Ε, και οι εργασίες του Dick Herring είδαν ότι υπάρχει τρόπος να μετρήσει κανείς ότι η κρίση των τραπεζών μπορούσε να έχει ε, αποφευθεί με πληροφορίες που είχε η αγορά 6 έως 12 μήνες νωρίτερα. Εάν λοιπόν θέλουμε να ανακτήσουμε την ρύθμιση των αγορών θα πρέπει να δώσουμε εις τους ρυθμιστές την εξουσία να ενεργήσουν διότι εάν ένας υπεύθυνος θέλει να επέμβει στην τράπεζα ακόμη και αν πρόκειται ε, να υπάρξει χρεοκοπίες θα χρησιμοποιηθούν όλα τα ένδικα μέσα για να αποφευθεί η έκβαση ενώ πρέπει να επιτρέψει κανείς τους ρυθμιστές αυτούς να επέμβουν παρέμβουν για να μην φτάσουμε στο χείλο του γκρεμού πρωτού φτάσουμε. Φτάσαμε στο τέλος του πρώτου γύρου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Γιόγκαν και σας ε, κύριε, σας ευχαριστούμε πολύ. the... Και τώρα θα καλέσω τους εισηγητές για το δεύτερο γύρο. Τον κύριο Μπέρμπερ και τον κύριο Κεβέ, παρακαλώ.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 Okay, Συνάδελφοι, περνάμε τώρα στο δεύτερο γύρο και για την <clears throat> διαθεσμική συνεργασία. Ένα θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Συζητήσαμε σε αυτήν την Κοινοβουλευτική Επιτροπή αυτό το θέμα ήδη αρκετές φορές. Γνωρίζουμε ότι Είχαμε ελπίσει κιόλα ότι όταν άρχισε η λέσχη των 20 τις συνεδριάσεις της και ξεκίνησαν με συστάσεις και τα λοιπά, ελπίζαμε ότι θα είμαστε σε θέση να προσκλεί, να συγκλίνουμε και ότι δεν θα υπήρχαν περαιτέρω αποκλήσεις. Πρέπει όμως να παραδεχθούμε, τουλάχιστον εγώ ίδιος και ομιλώ για τον εαυτό μου, έχω την εντύπωση που αποκόμισα ότι δεν είμαι βέβαιος, δεν είμαστε βέβαιοι ότι θα έχουμε μια πραγματικά συντονισμένη απάντηση σε σχέση με την κρίση στο τέλος τέλος και μπορεί να παρεκκλίνουμε προς διαφορετικές κατευθύνσεις. Αυτό θα ήταν κρίμα φυσικά γιατί θα άνοιγε πόρτα και παράθυρο για να υπάρχει ρυθμιστική δράση ε, προς ε, κάθε κατεύθυνση και με παρεκκλίνουσες δράσεις. Αλλά θέλω να δω από πλευράς των εισηγητών μήπως αυτό είναι ένας, μια ε, επιφανειακή αντιμετώπιση. Ξεκινάμε με την κυρία Μπερβουέλ που είναι <clears throat> επικεφαλής στο, για τις διατλαντικές σχέσεις και ε, μελέτες στο Ατλαντικό Συμβούλιο <clears throat> των ε, Ηνωμένων Πολιτειών στην Ουάσιγκτον. Και έχουμε και τον κύριο Κερέ, Γενικό Διευθυντή ε, που ε, σε σχέση με το Υπουργείο Οικονομικών στην ε, Γαλλία. Η κυρία Μπέρβολ είναι η πρώτη που θα παρέμβει. Έχετε τον λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Είναι χαρά να παρίσταμε εδώ ενώπιον σας και επίσης προσβλέπω επίσης στο να... Συγγνώμη μια στιγμή να το... Προσβλέπω επίσης στο... Εντάξει, ευχαριστώ. Ανθυμονώ να σας συναντήσω και στην Washington την επόμενη εβδομάδα. Θα μιλήσω γενικότερα κάπως Υπάρχει αυτή η πρόκληση όσον αφορά την Κοινοβουλευτική Επιτροπή. Μπορεί αυτή η Κοινοβουλευτική Επιτροπή αντιμετωπίζοντα την χρηματοοικονομική κρίση να συνεργαστεί με την Ουάσιγκτον και ιδιαίτερα με το Κογκρέσο με έναν τρόπο ώστε να θεσπιστεί ένα πρότυπο μια νέα συνεργασία μεταξύ τη Ευρωβουλή και του Κογκρέσου των Ηνωμένων Πολιτειών. Και αυτό που θέλω να επικεντρώσω την προσοχή μου είναι στο να δούμε τι μπορεί να γίνει στο μέλλον για την ε, τον πριτανεύοντα ρόλο της λειτουργικής αντιμετώπισης και όχι τόσο της τυπικής αντιμετώπισης. Αυτή η κρίση προσφέρει ευκαιρίες ε, παράλληλα με κινδύνους και θέλω να γίνει κατανοητό αυτό. Θα μιλήσω. γίνεται περισσότερος λόγος σε σχέση με τους κινδύνους και τις ευκαιρίες για το τι πρέπει να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και τι πρέπει να κάνει η Ευρωβουλή <clears throat> αντί το τι κάνουν ή πρέπει να κάνουν η ΙΠΑ. Αυτή είναι η ε, ενημέρωση που είχα για να επικεντρωθώ στο τι γίνεται σε σχέση με τις ΙΠΑ και θα πρέπει να είναι κατανοητό ότι οι παρατηρήσεις αυτές γίνονται από ένα άτομο που είναι φίλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Υπάρχουν θεμητέ ανησυχίες λοιπόν. Όλο και περισσότερες ε, πληροφορίες για το τι συμβαίνουν στην Ευρώπη, τι συνέβη στην Ευρώπη σε σχέση με το ευρώ. Έχουμε σχόλια για την αποσύνθεση, την διάλυση του ευρώ και είχαμε και ένα δημοσίευμα στο Washington Post για το τι Ποιε επιπτώσει μπορεί να έχει αυτό στην αμερικανική ε, ε, σημερινή συγκυρία σε σχέση με το, ε, τις προοπτικές. Και όλα αυτά ε, έχουν και τον κίνδυνο που συνεπάγονται της ε, διάβρωσης της ευρωπαϊκής αξιοπιστίας ε, και οικονομικά και πολιτικά. Αυτά όμως δίνουν ευκαιρίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρώτα απ' όλα να δείξει την ικανότητά της ότι είναι σε θέση η Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις η ίδια που είναι έχει ρόλο κλειδιού για να, ε, την αποκατάσταση της αξιοπιστίας απολοράσης. Αυτό που θέλω να κάνω είναι να επικεντρωθώ σε θέματα επί της ουσίας και επί της λειτουργικής τους επίπτωσης και όχι για τους μηχανισμούς. Οι μηχανισμοί είναι σημαντικοί. Υπάρχει μια ολόκληρη, ένα, ένας ολόκληρος περίγυρος ε, θα έλεγα ε, και έχουμε επικεντρωθεί σε αυτό αλλά πρέπει να αποκλίνουμε λίγο περισσότερο από αυτή την επικέντρωση και να δούμε για ποια θέματα κάνουμε λόγο επί της ουσίας. Υπάρχει μια εντύπωση στην Washington σήμερα, αντιμετωπίζοντας θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεγάλης απογοήτευσης. Δεν κατανοούν το πώς λειτουργεί η Ευρώπη σε αυτή την μεταβατική περίοδο μετά τη συνθήκη της Λισαβόνα. και δεν υπάρχει η δυνατότητα, πολλοί δεν έχουν την όρεξη καν να επενδύσουν στο να κατανοήσουν περισσότερο ή να εξοικειωθούν με πολλά πράγματα. Όμω αυτά έχουν τεράστια σημασία την Washington. Κάνοντας λόγο για αυτά θέλω να κάνω λόγο εν συντομία για το θεσμικό περίγυρο όσον αφορά και την ε, προηγούμενη κυβέρνηση Μπού και τη σημερινή Ομπάμα και για τις θεσμικές μεταρρυθμίσεις ε, όσον αφορά τις σχέσεις Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Κογκρέσου, Ευρωπαϊκής Ένωσης ΗΠΑ και ιδιαίτερα για ποια θέματα θα πρέπει να κάνουμε λόγο. Οι χρηματοοικονομικές ρυθμίσεις είναι ένα θέμα που έχει σημασία κλειδιού και πρέπει αυτό να βρίσκεται πάνω πάνω στην ημερησία διάταξη προτεραιότητα. Και η οικονομική διακυβέρνηση. Δεν θα κάνω μια εξαντλητική απαρίθμηση όσον αφορά τα θεσμικά θέματα. Πολλοί από εσά είσαστε πολύ καλά εξοικειωμένοι για τα ιστορικά αυτά θέματα. Είναι όμω πολύ ασυνήθιστη η, α το πω έτσι, ε, συγκυρία αυτών των στοιχείων υπό το αμερικανικό πρίσμα. Δεν έχουμε δομημένες και διαθρωμένε σχέσει όπω αυτέ με την Ευρώπη με άλλε χώρε. Μία εξαίρεση είναι η Κίνα πολύ πρόσφατα. Στρατηγικό οικονομικό διάλογο σε σχέση με αυτή τη χώρα. Την τελευταία εβδομάδα ε, ε, το Υπουργείο, από πλευρά Υπουργείου Οικονομία είχαμε επαφές με τους Κινέζους. Έχουμε ένα ε, περισσότερο θα έλεγα ρουτινιέρικο ε, πλαίσιο σχέσεων με τις άλλες χώρες. Όμως αυτό σε σχέση με την Ευρώπη έχουμε και την ε, Σύνοδο Κορυφής Ευρώπης Ρωσίας Παράλληλα με τις πολλές, τα πολλά θέματα στην διατλαντική ημερήσια διάταξη έχουμε και την ανάπτυξη θεματολογικά διαλόγων με άλλες χώρες. Μέσα σε ένα διαρθρωμένο πλαίσιο. Έχουμε ένα διάλογο για τη δικαιοσύνη, τον ε, διάλογο για τη ρύθμιση των αγορών, το διάλογο για τα θέματα ασφάλειας, έχουμε ε, διάλογο σε σχέση με τους ε, νομικούς επαείοντες και νομικούς συμβούλους, έχουμε το ΤΕΚ που ελπίζουμε ότι σύντομα θα ξαναξεκινήσει με νέα, ας το πω έτσι, τόνωση όσον αφορά το Ενεργειακό Συμβούλιο. Και σε σχέση και με τις δύο όχθες του Ατλαντικού είναι αναγκαία αυτή η ε, προσέγγιση. Μπορεί να αλλάζει ε, ανακυκλούμενα μέσα στον χρόνο η επικέντρωση. Όμως ε, αυτή είναι, θα έλεγα, η σωστή προσέγγιση. Πρέπει να υπάρχει ένας διαθρωμένος διάλογος. Σύνοδοι κορυφής. Όλοι μπορούμε να συνάγουμε το συμπέρασμα ότι είχαν ένα θετικό αποτέλεσμα και υπάρχουν